Αναλαμβάνεται η συνεδρίασή μας ε, που διεκόπη στις 13 Φεβρουαρίου, 3 Φεβρουαρίου συγγνώμη, 2011. Τα πρακτικά έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Υπάρχουν σχόλια. Παρατηρήσεις σε σχέση με τα πρακτικά ή τα κείμενα. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις για τα πρακτικά, οπότε υιοθετούνται τα πρακτικά. Έχω να σας πω τα εξής σε σχέση με την ε, επανάληψη τη.